Colleagues, um, if you could please take your places. Mr. Becker. Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι. Κύριε Μπέκερ. That would be appropriate. okay, colleagues, settle down. Thank you. Um, okay, colleagues, thank you. Ευχαριστώ συνάδελφοι που ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση και θα ήθελα να καλωσορίσω τη Ιωάννα Μίκη Λάιτνερ για το πρώτο σημείο της ημέρησης διάταξης, την ε, Ομοσπονδιακή Αυστριακή Υπουργό Εσωτερικών. Θα έχουμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων, γιατί τον η Αυστρία ανέλαβε το Σεπτέμβριο μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουμε την τραγική κατεπίγουσα ανθρωπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζουν χώρες ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταιγισμό των προσφύγων. Η πρωτοβουλία λέγεται Save Lives, ε, σώζουμε ζωές. Και ήρθε εδώ για να μας παρουσιάσει την πρωτοβουλία και να συζητήσει με τους ευρωβουλευτές. Επίσης έχουμε και την διάσκεψη δωρητών σε υπουργικό επίπεδο που οργανώνει η Πατία Αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων και θα γίνει σε 9 Δεκεμβρίου στη Γενέβη. Εκεί οι χώρες ε, θα υποσχεθούν δωρεές για να αντιμετωπιστεί το κύμα σύρων προσφύγων και επίσης στην επόμενη συνεδρίαση θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για το Φόρουμ Επανεγκατάστασης και Επανατοποθέτησης. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε στην Επιτροπή μας έναν Υπουργό που αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία που μας ενδιαφέρει, γιατί το θέμα της επανεγκατάστασης, όπως ξέρετε κυρία Υπουργέ, είναι ένα ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέτοιες πρωτοβουλίες. Γι' αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία που αναλάβετε σε υπουργικό επίπεδο και προωθείτε στα κράτη-μέλη. Θα συζητήσουμε τη δική σας εμπειρία και θα σας ε, ενημερώσουμε και για τις δικές μας. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα καλά λόγια με τα οποία με υποδεχτήκατε. Χαίρομαι που με έχετε προσκαλέσει εδώ στην Επιτροπή σας ΛΥΜΠΕ. Με ενδιαφέρει όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο η συνεργασία με τα κοινοβούλια, αλλά βεβαίω και στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που σήμερα μπορώ να σας παρουσιάσω και αναπτύξω την αυστριακή μας πρωτοβουλία Save Lives. Γνωρίζετε όλες και όλοι ότι αντιμετωπίζουμε εντελώς έκτακτες καταστάσεις και τέτοιες έκτακτες καταστάσεις χρειάζονται επαγγελματικέ και ταχύτατες λύσεις. επαγγελματικέ και ταχύτατες ιδίως όταν εξετάζει κανείς τα σημαντικά ρεύματα μετανάστευσης και όταν γνωρίζουμε ότι στις γειτονικές χώρες της Συρίας πραγματικά δεν χωράνε πλέον τα στρατόπεδα προσφύγων τον κόσμο. Και έχουμε βέβαια και την Βόρεια Αφρική, όπου χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να περάσουν απέναντι. Ταυτόχρονα έχουμε και την άλλη θεματική, ότι δηλαδή ειδικώ στην Ευρώπη εν μέρη είναι υπερβολικά επιβαρημένα τα εθνικά συστήματα ασφαλίσεων. Δέκα δηλαδή από τις 28 χώρες μέλη δέχονται το 90% των αιτήσεων ασύλου. Ειδικώ λοιπόν στις ιδιαίτερα επιβαρημένες χώρες η αντιμετώπιση ε, δεν μπορεί να είναι βέλτιστη. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου απαιτούνται μέτρα σε δύο επίπεδα. Αφενός χρειάζεται να θεσπιστεί μια διαδικασία που να επιτρέψει την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και βεβαίως και των ε, παράνομων διακινητών, από την άλλη μεριά πρέπει να προσφέρουμε νόμιμους δρόμους ασφαλούς έλευση στην Ευρώπη για τους νόμιμους μετανάστες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, ο στόχος του Project Save Lives. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φροντίσουμε τους πρόσφυγες εκεί και να πάμε να βρούμε εκεί όπου βρίσκονται, ώστε να μην πέσουν βορρά των διακινητών. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε επαγγελματίες αξιόπιστους εταίρους όπως τον ε, είπα το αρμοστή των Ηνωμένων για τους πρόσφυγες. Η πρωτοβουλία πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύνολο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται βεβαίως η υποστήριξη και συμμετοχή όλων των χωρών μελών σύμφωνα με μια κλίδα ισοδίκης κατανομής στο πνεύμα της αλληλεγγύης, διότι η αλληλεγγύη βεβαίως είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά λοιπόν στο θέμα αυτό του ασύλου των ροών μεταναστών η Ευρώπη μπορεί να θρηματιστεί αν δεν βρει καινής λύση. Άρα πρέπει η προσέγγιση μας να είναι κοινή, κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για να προσφέρουμε λύσεις και βοήθεια. Πρέπει να τονίσω πρώτα ότι εδώ χρειάζεται, όπως είπα, μια κλίδα ισοδίκης κατανομής μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι αυτή η ισοδίκη κατανομή δεν υπάρχει ακόμη, θα πρέπει ακόμη να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Θα χρειαστούμε την βοήθεια του ΕΑΣ και άλλων οργανισμών. Δεύτερο, το δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι βεβαίως η υποδοχή των προσώπων που έχουν ανάγκη προστασίας εδώ στην Ευρώπη σύμφωνα με αυτή την κλίδα κατανομής. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος πιέζει. Ιδιαίτερα στις ζώνες όπου σημειώνονται συγκρούσεις τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα από τη Βόρεια Αφρική μέχρι την Εγγύς Ανατολή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επαγγελματική προεργασία βεβαίως αλλά κυρίως πρέπει αυτή να είναι ταχύτατη. Γνωρίζω ότι χρειάζεται και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο του χώρα μέλου, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά βέβαια και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό προσέρχομαι ενώπιόν σας για να παρακαλέσω να μας χορηγήσετε την υποστήριξη αυτή. Ως πολιτικοί θύνοντες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς οι διακινητές στέλνουν στον όλεθρο όλο και περισσότερους ανθρώπους. Όλοι έχουμε μπροστά μας έντονες τις εικόνες όταν σκεφτούμε ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες ολόκληρες χιλιάδες ανθρώπων χάθηκαν στα κύματα της Μεσογείου. Πρέπει να τους προστατεύσουμε απέναντι στους διακινητές. Ταυτόχρονα, όπως είπα, πρέπει να προσφέρουμε νόμιμους, ασφαλείς δρόμους προς την Ευρώπη για εκείνους που είναι νόμιμοι μετανάστες. Έτσι ώστε να αφαιρέσουμε την πίεση κιόλας από τα εξωτερικά ε, σύνορα και επίσης από τα συστήματα υποδοχής. Αυτή λοιπόν η δική μας αυστριακή πρωτοβουλία Save Lives υποβάλλει μια συγκεκριμένη πρόταση και χαίρομαι που σήμερα μάλιστα μπόρεσα να συζητήσω με τον νέον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα του υποβάλω την πρόταση, πρόταση που προβλέπει την συμμετοχή όλων των χωρών μελών και όπως είπα δίκαιη κατανομή των ε, μεταναστών. Με την πρόταση αυτή, λοιπόν, πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποφύγουμε οι άνθρωποι αυτοί να περνούν με περιπετειώδη τρόπο τη Μεσόγειο και να ρισκάρουν την ίδια τη ζωή. Και με την πρόταση αυτή έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αφαιρέσουμε το γόνιμο έδαφος κάτω από τα πόδια των διακινητών. Μπορεί να γίνει αυτό, ιδίως αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια δίκαιη ισοκατανομή των μεταναστών στις διάφορες χώρες μέλη. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας, η Επιτροπή των Θεμελιδών Ελευθεριών, που δέχεται να αρχίσει τη συζήτηση αυτή μαζί μας. Εμείς έχουμε αποφασίσει να προωθήσουμε το έργο μας αυτό, το project μας αυτό και να το συζητήσουμε σε όλα τα επίπεδα, το εθνικό, το ευρωπαϊκό, για να καταλήξουμε σε μια ανθρώπινη και ανθρωπιστική λύση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Είναι καλό που ακούσαμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι καλό να έχουμε επαφές με υπουργούς που κινούνται σε αυτό το τομέα. Είναι καλό για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πήρατε το χρόνο να έρθετε εδώ. Τώρα ο λόγος πηγαίνει στα μέλη μας. Δύο από τα μέλη μας από την Αυστρία. Ο κύριος Μπέκερ και κύριος Ο κύριος Μπέκερ πρώτος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης που μας προσφέρατε αυτή την ευκαιρία ενημερώσεως. Εσείς κύριε Υπουργέ, αγαπητή Άννη, εσάς σας ευχαριστώ για αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται πραγματικά στο κέντρο όλων των ανησυχιών μας. Κυρίως αν σκεφτούμε την ανάγκη να φανούμε αλληλέγγυοι και ταυτόχρονα με αποφασιστικό τρόπο να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση. Είναι σημαντικό εμείς οι Ευρωπαίοι σε αυτήν την κρίση που αντιμετωπίζουμε να παραμείνουμε ενωμένοι. Η πρότασή σας είναι πραγματικά σημαντική συμβολή για την ενότητα αυτή έχουμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε την παράνομη εγκληματική δραστηριότητα των διακινητών, ταυτόχρονα οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας για την προστασία των ανθρώπων. Και εδώ είναι παραδειγματική φύσεως η πρωτοβουλία Έχω ερωτήσει που θα ήθελα να σα υποβάλω σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος στην Επιτροπή μας. Η μία ερώτησή μου αναφέρεται στο πώς τίθεται το πρόβλημα. Εάν θεωρήσουμε ότι στο πρόγραμμά σας αυτό, Save Lives, περιέχεται ήδη και παίζει ένα σημαντικό ρόλο η κλίδα κατανομής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στη μελλοντική ρύθμιση της μετανάστευσης και ιδίως της παράνομης μετανάστευσης, η κρίδα που προτείνεται τώρα αποτελεί ας πούμε το βασικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα καταλήξουμε να αναπτύξουμε την τελική κλίδα. Δεύτερο, πώς φαντάζεσαι αγαπητή Άννη την παραπέρα εξέλιξη του συστήματος του Δουβλίνου. Αυτό είναι κέρια σημασίας. Και τρίτο, πώς βλέπεις από τη δική σου σκοπιά της Ομοσπονδιακής Υπουργού την στήριξη που μπορεί να προσφέρει το Συμβούλιο. Τέλος, θα εκφράσω μια ελπίδα. Η Επιτροπή Λίμπε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή, όπως το έχουμε συνηθίσει εδώ, διακομματικά, από όλες δηλαδή τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Ο κύριος Βάιντεν Χόζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Κλοντ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ εγκαρδίως που προσήλθατε εδώ ενώπιόν μας. Συγκαταλέγω μεταξύ εκείνων που σας ασκούν και κριτική και που σε ορισμένα πράγματα έχουμε διαφορετική άποψη από εσά. Είχα την εντύπωση μάλιστα ότι το καλοκαίρι ξέφυγε η συζήτηση διότι καταλήξαμε να μιλούμε μοναχά για κλείσιμο συνόρων και άλλα σχετικά. Σας διαβεβαιώ όμως ότι σήμερα αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος από την πρωτοβουλία σας. διότι συμβάλλεται στο να ξεφύγουμε λίγο από το παιχνίδι εκείνο που λέει ότι πάντα φταίει ο άλλος, ο οποίος δεν φροντίζει να ε, ασφαλίσει τα σύνορά του και το καθεξής. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία σας είναι σημαντική για δύο λόγους. Αφετέρου, αφενός μάλλον, διότι θεωρεί ότι προφανώς δεν είναι δυνατόν να είμαι υποχρεωμένο να υποβάλω την αίτηση ασύλου μου όταν φτάσω στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτός είναι ο λόγος που αναγκάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους να περνούν τη Μεσόγειο για να έρθουν εδώ. Εάν μετατεθεί η διαδικασία αυτή αλλού, αυτό θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική διέξοδο από αυτή την αδιέξοδη κατάσταση. Το συζητήσαμε αυτό σήμερα το πρωί. Ποιε δυνατότητε ενδεχομένω θα υπήρχαν να προσφερθούν άλλες τέτοιες πρόσθετες δυνατότητες εισόδου και οφείλουμε να καθίσουμε να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Όχι απαραίτητα να συνεννοηθούμε μονάχα με τον UNHCR, αλλά να δούμε και τι μπορούν να κάνουν οι πρεσβευτές, οι, πρεσ, οι πρεσβείες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι αυστριακές πρεσβείες κάποτε είχαν τη δυνατότητα να δίνουν ειδικέ θεωρήσεις για τέτοιες περιπτώσεις ασύλου. Και αυτό είχε βοηθήσει σε μια χαλάρωση της καταστάσεως. Χαίρομαι λοιπόν που για πρώτη φορά βλέπω να μελετώνται και κάποιες άλλες δυνατότητες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι βεβαίως αυτή η κλίδα κατανομής είναι απόλυτα λογικό και σκόπιμο να ζητήσουμε να κατανέμονται σε όλες τις χώρες μέλη. Θα δούμε πώς θα γίνει βέβαια γιατί είναι και άλλες πτυχές του ζητήματος όπως επανένωση οικογενειών κλπ. Αλλά ασφαλώς είναι σκόπιμο και χρήσιμο να κατανεμηθεί το βάρος σε όλες τις χώρες μέλη. Και να ξεφύγουμε λίγο και από αυτό το στενό σύστημα του Δουβλίνου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν συμφωνείτε ότι καταρχήν πρέπει αυτό να σκεφτούμε. Να αντικαταστήσουμε ίσως με κάτι άλλο το σύστημα, το σύστημα του Δουβλίνου. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει βεβαίως από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά κάπου νομίζω αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο για πολλούς από εμά ότι το Δουβλίνο δεν λειτουργεί. Εφόσον βέβαια δεν διαθέτουμε τίποτε άλλο, ασφαλώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό παρόλες τις ελλείψεις του. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Χαίρομαι επίσης που επιλέξατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τον τόπο όπου θα παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Αυτό νομίζω είναι ένα δείγμα σεβασμού το οποίο δέχομαι απολύτως ως δείγμα σεβασμού προς τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την τελευταία δήλωση. Η κυρία Σιρεβέλ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στην Υπουργό και σας καλωσορίσω που ήρθατε εδώ σήμερα για να παρουσιάσετε τη σημαντική πρωτοβουλία. Είναι πάντα σημαντικό για μας να μπορούμε να ακούμε και να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές, είτε από κράτη-μέλη, είτε από εμπειρογνώμονες, είτε από διάφορους άλλους φορείς. Εκτιμώ το ότι υπογραμμίζεται την απελπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζουν μετανάστες. Πολύ συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να θέσουν τη ζωή τους στα χέρια των διακινητών. Τους λείπουν οι δυνατότητες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς και νομίμως. Δεν θα δούμε λύση όσον αφορά τους θανάτους στη Μεσόγειο, όσον αυτή είναι η μόνη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την πρωτοβουλία που παρουσιάσατε εσείς από την Αυστρία. Συμφωνώ μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής φέρουν τεράστια ευθύνη όσον αφορά τι διεθνεί ανθρωπιστικέ προσπάθειε. Καλωσορίζω την πρότασή σα για εφαρμογή κοινή ευρωπαϊκή ε, προσπάθεια διευθέτηση μαζί με την ύπατη αρμοστία. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να δράζεται επί της αρχής της αλληλεγγύης και να υπάρχει ευρωπαϊκή ε, κοινή υποχρέωση για τη μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση. Μόνο λίγα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτή τη ε, διαδικασία επανεγκατάστασης και μερικά από τα κράτη δέχονται μόνο περίπου μέχρι 100 άτομα το χρόνο. Ε, δεν είναι τίποτα το πρόγραμμα, ούτε καν αγώνα στον ωκεανό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάσταση μεταναστών. Αν το δει κανεί στο διεθνέ προσκήνιο, μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα. Ταυτόχρονα να αυξήσουμε την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013 μόνο τρία κράτη-μέλη δέχτηκαν 57% όλων των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτιώσεων. Αν εισάγουμε ένα είδος κλίδας κατανομής ή σύστημα ποσοστώσεων μεταξύ κρατών μελών, αυτό θα είναι πολύ κρίσιμο. Ε, θα πρέπει να βασίζεται επί ποσοτικών στοιχείων όπως το ΑΕΠ της χώρας, πληθυσμός, μέγεθος της επικράτειας της χώρας κλπ. Ακόμα πιο σημαντικό, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα ποιοτικά στοιχεία, όπως οικογενειακές σχέσεις, διαδικασίες, προοπτικές ένταξης στη χώρα, ε, γνώσεις γλωσσών κλπ. Αν δεν λάβουμε υπόψη τα ποιοτικά αυτά στοιχεία, τότε θα δημιουργηθούν προβλήματα για την ένταξή του κάτι που δεν χρειάζεται και το σύστημα ποσοστώσεως θα πρέπει να επιδιώκει ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών, χωρί όμω αυτό να γίνεται υποχρεωτικό, δηλαδή να πρέπει να πάει ο ετών άσυλο σε συγκεκριμένη χώρα για να υποβάλει την αίτησή του. Πρώτη ερώτηση. Προβλέπετε ίσω ένα σύστημα ποσοστώσεων ή κλίδα κατανομής που θα είναι υποχρεωτικά ή εθελοντικά για τον ετώντα άσυλων. Ε, πόση ευελιξία θα υπάρχει τα ποιοτικά στοιχεία κατά πόσο θα λαμβάνονται υπόψη, ενώ θα είναι υποχρεωτικό ταυτόχρονα για τα κράτη-μέλη να ε, αναλάβουν το μερίδιο των ευθυνών τους. Δεύτερο ερώτημα. Η πρότασή σας πώς έγινε δεκτή στο Συμβούλιο, πώς τη δέχτηκαν τα άλλα κράτη-μέλη, υπάρχει αρκετή υποστήριξη να προχωρήσουμε με αυτές τις ιδέες. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ συχνά εμείς αυτή την Επιτροπή θα θέλαμε να είμαστε μια μίγα εκεί και να ακούμε τι λένε οι άλλοι. Εσείς έχετε μια υπέροχη δυνατότητα να ανταλλάξετε τις εμπειρίες σας ε, που έχετε στο Συμβούλιο και να μας πείτε τι γίνεται εκεί. Μετά, ξέρετε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το στάδιο θα ήταν έτοιμη ή σύντομα θα ήταν έτοιμη να επεξεργαστεί και να μας υποβάλει πιλωτικό πρόγραμμα με αυτά τα στοιχεία μέσα. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, Έχετε κάποιες ενδείξεις πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σεσίλια. Κυρία Υπουργέ, σίγουρα θα χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία να μας πείτε τι λένε οι συναδελφοί σας στο Συμβούλιο. Συνάντησα τον ομόλογό σας στο Γερμανό πριν από μία ώρα. Μπορώ να συγκρίνω, υπάρχει αντίθεση μεταξύ σας. Τέλος πάντων. Είναι πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις, άρα βλέπετε πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτό το θέμα εδώ και πόσο εκτιμούμε όταν ακούμε αυτά τα παραδείγματα που μας Ο κ. Τζοφσκι, ο Τόμας Τζοφσκι είναι επόμενος. Έχει το λόγο, Τόμας. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ανάλυση, καθώς και για την πρωτοβουλία σας που ε, μας παρουσιάσατε. Εγώ όμως δεν είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής, διότι βλέπω πολλές, πολλά προβλήματα να έχει αυτή η πρωτοβουλία. θέμα που στη Γαλλία πολλά εθνικιστικά κόμματα αλλά και σε άλλες χώρες το θέτουν ως μέγα πρόβλημα. Τα ποσοστά, οι ποσοστώσεις, καλύτερα, αποτελούν το κόκκινο πανί για όλους εκείνους που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω όμως και ερωτήσει τώρα που καλύτερα σας τις πω στα τσεχικά γιατί είναι πιο εύκολα για μένα. Μέχρι τώρα μίλησα γερμανικά. Συνήθως είμαι υπέρ της Αυστρίας και χαίρομαι πολύ που το θέτει το θέμα η Αυστρία. Θα συνεχίσω όπως είπα τώρα στα τσεχικά. Έλεγα λοιπόν ότι κοιτάξτε, εάν οι μετανάστες ή αυτοί που ζητούν άσυλο δεν διέλθουν ολόκληρη την διαδικασία Υποβολή Πού θα επιστραφούν, αυτή είναι η ερώτηση που θέτουν όλοι στην τσεχική δημοκρατία. Μετά το ζήτημα των ποσοστώσεων. Η τσεχική δημοκρατία δεν έχει μείζον πρόβλημα με το ενδεχόμενο υποδοχής μεταναστών. Θα γίνει μετά όμω. Πώς θα προχωρήσει η διαδικασία ενσωμάτωση. Θα μάθουν τα τσεχικά για παράδειγμα. Είδατε ο ίδιος ο πρόεδρος πώς προφέρει το όνομά μου δεν τα καταφέρνει γιατί η γλώσσα μας είναι πιο δύσκολη στην Ευρώπη. Εμείς οι Τσέχοι λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι θα καταφέρει κανένας μετανάστης ποτέ να μάθει τσεχικά. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ίσως κάποιοι άλλοι, Σλοβάκοι ή Ουκρανοί, να είναι πιο εύκολο να δεχτούν μετανάστες από σλαβικές χώρες. Αλλά εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν. Εγώ έχω πάει και έχω επισκεφθεί μετανάστες από την Βυρμανία και από αλλού και αυτοί δεν κατάφεραν να ενταχθούν καθόλου. Δεν μπορούν να μάθουν τα τσεχικά δεν είναι σαν τα αγγλικά τα γαλλικά. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά έχω και μια άλλη ερώτηση. Ίσως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα καλύτερα σε εθελοντική βάση. Κάθε χώρα μέλος δηλαδή η ίδια να κρίνει αν επιθυμεί να υποδεχθεί κάποιον αριθμό μεταναστών σε εθελοντική βάση. Είχα πάει σε ένα συνέδριο στην Ιταλία και βγήκαν μερικοί και είπαν ότι επί του παρόντος οι ποσοστώσεις δεν αποτελούν λύση. Ακούσατε και τους συναδέλφους της Σικελίας που έρχονται και διορθώνουν τα νούμερα που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι φαίνεται πως είχαμε εσφαλμένα στατιστικά δεδομένα Δηλαδή κάποιοι μιλούν εδώ για εκατοντάδε μετανάστε, ενώ πρόκειται για λίγε δωδεκάδες. Πώ θα αντιμετωπίσει όμω το πρόβλημα η ε, Ένωση και πού θα βρει τη χρηματοδότηση. Τέτοια ερωτήματα με απασχολούν. Εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι το ίδιο αισιόδοξο όπω ο συνάδελφό μου Μπέκερ, αλλά έχω πάρα πολλέ ερωτήσει και πολύ λίγε απαντήσει. Ευχαριστώ. Τελευταία που θα πάρει το λόγο είναι η Helga Stevens. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επανεγκατάσταση των προσφύγων. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποσκοπούμε στη βοήθεια, να αποβλέπουμε στη βοήθεια των προσφύγων, των όσων τουλάχιστον προσφύγων χρήζουν προστασίας. Πώς όμως θα τα καταφέρουμε. Κανονικά ισχύουν οι κανόνες του Δουβλίνου. Οπότε υποβάλλεται η αίτηση ασύλου στο πρώτο κράτος φτάνει ο Πώς θα γίνει κατόπιν η, η κατανομή με βάση την κλίδα κατανομής. Αυτά δεν τα πολύ κατάλαβα. Συνάδελφοι, εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ε, παρεμβάσεων. Κυρία Υπουργέ, αν είσαστε έτοιμοι, τέθησαν ουσιαστικά ζητήματα. Σας παρακαλώ, απαντήστε. Äh, Είμαι στη διάθεσή σας και πρόθυμη να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Η δυσκολότερη πρόκληση δεν είναι η γενική πρόταση, το γενικό πλαίσιο, αλλά οι λεπτομέρειες και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η πρωτοβουλία αυτή σε διάφορα επίπεδα. Όπως είπε η βουλευτής από τη Μεγάλη Βρετανία, θα, θα πρέπει να ξεχνούμε πόσο απεγνωσμένοι, πόσο απελπισμένοι είναι οι πρόσφυγες, σε τι απόγνωση βρίσκονται. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι διώκονται στη χώρα τους, φοβούνται ότι θα χάσουν τη ζωή τους, ότι θα γίνουν θύματα βιασμού. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή εδράζεται πάνω απ' όλα στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες φυσικά κάνοντας τη διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Και είναι λογικό κάποιοι μετανάστες να χρειαστεί να επαναπατριστούν. Αναφέρθηκε και η διαδικασία μέσω των προξενείων και των πρεσβειών. Φυσικά θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με εταίρες μας που έχουν πείρα στο θέμα αυτό, όπως είναι η πατιαρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ε, άνθρωποι με πείρα και επαγγελματίε θα κρίνουν αν ε, ο μετανάστευς πραγματικά χρήζει προστασία ή όχι. Γιατί δεν θα εφαρμόσουμε την κλίδα κατανομής για πρόσφυγες που δεν χρήζουν προστασίας, αλλά μόνο για ανθρώπους που πραγματικά διώκονται και κινδυνεύει η ζωή τους. Και με βάση την κλίδα αυτή κατανομής ε, θα παραπέμπονται οι πρόσφυγες στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και θα εξετάζονται οι αιτήσει τους. Υπάρχουν φυσικά και μεταβατικές λύσεις. Μπορεί κανείς να έρχεται απευθείας στην Ευρώπη και να καταθέτει απευθείας ε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα το αίτημά του για άσυλο. Όμως στο μέλλον ο κανόνας θα είναι οι αιτήσει ασύλου να επί επιτόπου στις χώρες τους ενδεχομένως και σύμφωνα με τους κανόνες ή στα γραφεία του ε, είπα του αρμοστή και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία τότε να προσφέρουμε νόμιμες οδούς ασφαλείς οδούς στους ε, πρόσφυγες ώστε να μην αναλαμβάνουν το ρίσκο του ταξιδιού, το ρίσκο της φυγής και τελικά να μην πέφτουν θύματα των διακινητών. Αυτή είναι η συνολική ιδέα. Βεβαίως γνωρίζω ότι θα υπάρξουν μεταβατικές φάσεις όπου θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο να συμμετάσχουν εθελοντές. Επανέρχομαι στα όσα είπε ο συνάδελφός σας από την Τσεχία. Εγώ μεγάλωσα στα τσεχικά σύνορα. Είμαι παιδί δηλαδή παραμεθόριας περιοχής και γνωρίζω ότι η κατάσταση της Τσεχία είναι θαυμάσια και όταν κοιτάζω τις στατιστικές σας βλέπω ότι η Αυστρία σε χίλιους κατοίκους έχει δύο αιτήσει ασύλου, ενώ η Τσεχία σε χίλιους κατοίκους έχει 0,02. Η ασφάλεια, ωστόσο, για τον πρόσφυγα είναι το ίδιο καλή στην Αυστρία όπως είναι στην Τσεχία. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση και σε άλλες χώρες μέλη για να συμμετάσχουν ή ενδεχομένως να δηλώσουν διάθεση συμμετοχής σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Χώρες τέτοιες που μέχρι τώρα έχουν υποδεχθεί πολύ λίγους πρόσφυγες πολέμου. Έρχομαι λίγο τώρα και στο πρόβλημα της ενσωμάτωσης. Είναι κρίσιμο εφόσον έχει γίνει δεκτή καταρχήν η αίτηση ασύλου, να μπορεί να γίνει η ένταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου θα επανέλθει η ειρήνη στις πατρίδες τους, γνωρίζουμε ότι πολλοί θα θέλουν να επιστρέψουν εκεί. Βέβαια, πολλοί θα θέλουν να παραμείνουν. Αν ε, θυμηθώ για παράδειγμα τους Σύρους πρόσφυγες, το βλέπω αυτό. Και εκεί είναι απαραίτητο οι πρόσφυγες που θα παραμείνουν παροιμήν σε εμά δηλαδή ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να μπορούν να ενταχθούν. Και θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι και αυτοί βεβαίως να συνεργαστούν και να μάθουν και τις γλώσσες μας. Το κρίσιμο πάντως είναι να μπορούμε να προσφέρουμε μέτρα ένταξης και τα μέτρα αυτά βεβαίως θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τους ίδιους. Το να μάθουν μια ξένη γλώσσα πάντα είναι δύσκολο. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι ιδίω οι Σύριοι πρόσφυγες που συχνά είναι και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και έχουν και έφεση για την εκμάθηση γλωσσών είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουν να μάθουν τα τσέχικα πολύ γρήγορα και εύκολα. Εγώ πάντως σήμερα θα συζητήσω, σήμερα θα συζητήσω ακόμη με τον Επίτροπο. Θα τον αναπτύξω το πρόγραμμα ως μια ιδέα συνολικής ευρωπαϊκής λύσης με ειδική στόχευση σε αυτήν την συστηματική των ποσοστώσεων που θα πρέπει να είναι δεσμευτική για όλους. Γιατί τώρα ειδικά όπου έχουμε συμφωνήσει ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα ασύλου και επομένω όλοι θα έχουν κάποιε υποχρώσεις, πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των υποχρεωτικών ποσοστώσεων. Και στην Αυστρία έχουμε παρόμοιο πρόβλημα. Και εκεί βλέπουμε αυτή την ανισοκατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε την ανισοκατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βλέπουμε και στην Αυστρία. Μέρος των ομοσπονδιακών κρατηδίων μας εκπληρούν τις ποσοστώσεις τους, άλλο, άλλο μέρος όχι. Το ίδιο βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ απευθύνουμε ωστόσο έκκληση στην αλληλεγγύη σας. Και όπως είπα προηγουμένως, η ανισοκατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγκυται στο ότι 10 από τις 28 χώρες μέλη δέχονται και χειρίζονται το 90% των αιτήσεων ασύλου. Προτείνουμε τώρα λοιπόν η εξέταση των αιτήσεων ασύλου να γίνει στην τρίτη χώρα και μετά να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι δύσκολη η κατάσταση και γεμάτη προκλήσεις. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στον δρόμο της φυγής προσπαθούν να ξεφύγουν τον βιασμό, το, την τρομοκρατία, τη, τους φόνους. Είμαι βεβαίως στην διάθεση για να, συζητήσουμε, διότι υπάρχουν για την κατανομή διάφορα κριτήρια, όπως ο αριθμός των ε, του πληθυσμού και λοιπά. Το κρίσιμο εν προκειμένου είναι να αναλάβουμε να πούμε, τη δέσμευση να πούμε ναι για το πρόγραμμα. Είμαι βεβαίω ότι κανείς δεν έχει το συμφέρον να δει να αποτυγχάνει η Ευρώπη σε αυτό το σημαντικό θέμα. Γι' αυτό όπως είπα από την αρχή η Ευρώπη χρειάζεται επαγγελματικές λύσεις αλλά ταχύες λύσεις και γι' αυτό απευθύνω και πάλι έκκληση προς όλους και όλους να συμβάλλετε. Α, ξέχασα να απαντήσω σε μια ερώτηση για το Δουβλίνο. Εάν όντω το σύστημα αυτό εξεταζόμενο συνολικά αποδείξει ότι λειτουργεί, μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον αποδείξει εννοεί ότι δεν λειτουργεί. Μπορούμε τελικώς να το καταλήψουμε, αλλά χρειάζεται ω τουλάχιστον μεταβατική λύση το σύστημα του Δουβλίνου, έστω και από τροποποιημένη μορφή του. Και εφόσον υπάρξει σύστημα ποσοστώσεων που να εξασφαλίζει κάποια δίκαιη κατανομή, τότε νομίζω ότι όντω μπορούμε να εγκαταλείψουμε το σύστημα του Δουβλίνου. Αν δηλαδή υπάρξει μια δίκαιη κατανομή, δίκαιη ποσόστοση και αν αυτή τηρείται από όλου, τότε δεν θα χρειαζόμαστε εν τέλει το Δουβλίνο. Αυτό όμως θα είναι και το απότερο τέλος της διαδρομής. Περί αυτού πρόκειται. Σας ευχαριστώ και πάλι που μου προσφέρατε την ευκαιρία να αναπτύξω το πρόγραμμά μας ενώπιόν σας και επιτρέψτε μου μια ευχή ή μια παράκληση προς εσάς. Διαφημίστε το πρόγραμμα μας στους και στις συναδέλφους σας, αν μπορώ να το πω έτσι. Κάντε του διαφήμιση, ώστε όσο πιο πολύ να το δεχτούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ακούω τσεχική δυρμηνία στα αυτιά μου. Τι είναι, με τιμωρεί ο Θεός επειδή δεν προφέρω καλά το, τα τσεχικά ονόματα. Α, όχι, συγγνώμη, λάθος έγινε. Ένα τεχνικό πρόβλημα. Είπατε ότι καλό θα ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ένα εύρυθμο σύστημα ασύλου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει έργο, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν διατάξεις και υπάρχουν πρωτοβουλίες. Φυσικά έχουν αδυναμίες, τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά Σίγουρα όταν τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε ε, βοηθάνε και εμά. Γιατί αυτό που φοβόμαστε είναι ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι διατάξει που ήδη εγκρίνουμε. Γιατί η επανεγκατάσταση είναι ένα καλό παράδειγμα ε, των λεγόμενων μου. Όπω ε, είπε και η συνάδελφο, έχουμε άνηση εφαρμογή, τεράστιε διαφορέ και ανισότητε στην εφαρμογή τη πολιτική επανεγκατάσταση. Και υπάρχει και το θέμα των πολιτικών μα. Γιατί όσο πιο στενέ επαφέ έχουμε με το Συμβούλιο, τόσο το καλύτερο γιατί οι κύριοι συνομιλητές μας στην ε, μεταναστευτική πολιτική και πολιτική του ασύλου είναι τα μέλη του Συμβουλίου, γιατί τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτά που ψηφίζουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως είπατε θα πρέπει να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα και να προβάλλουμε, να διαφημίσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και για την συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ.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 Colleagues, Ναι και είμαστε όλοι παρόντες. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Όσοι είναι εδώ οι συνάδελφοι και το εκτιμώ ιδιαίτερο γιατί μείνατε πολύ πέμπτη απόγευμα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στη Frontex. Περνάμε στο σημείο 20, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί φαντάζομαι όλοι βιαζόμαστε να τελειώνουμε νωρί Είναι και πέμπτη απόγευμα. Για τη Frontex. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή, με τον εκτελεστικό διευθυντή μάλλον της Frontex. Τον περιμένουμε να πάσα στιγμή.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 that. So, um, Φυσικά υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για τον Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησικής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών. Ε, ζήτησα συγγνώμη από τον κύριο Λετζέρη που βάλαμε το θέμα αυτό πέμπτη απόγευμα, αλλά χαίρομαι γιατί πολλοί συνάδελφοι παρέμειναν για να ακούσουν την παρέμβαση του κυρίου Λετζέρη. Στις 26 Νοεμβρίου, πριν από μία εβδομάδα και με βάση με πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επελέγει ο κύριος Φαμπρίτσε Λετζέρη για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Frontex και δεδομένη στις μεγάλη σημασία που θα έχει η μελλοντική μα συνεργασία με τον εκτελεστικό διευθυντή, κρίναμε σκόπιμη τη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Όπω ε, είδαμε και στην ανακοίνωση για την καινή θέση, πριν ε, το διορισμό ο υποψήφιος ε, ε, μπορεί να δεχτεί πρόσκληση από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ακρόαση και μετά της ε, δηλώσεις του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υθετήσει γνωμοδότηση με τις απόψεις του για τον επιλεγμένο υποψήφιο. Κύριε Λετζέρη, έχετε το λόγο. Thank you Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι προσκεκλημένος Επιτροπής Πολιτικών Ελευθερίων Ανταλλαγή Απόψεων στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την εκλογή μου σαν εκτελεστικού διευθυντού του Frontex. Θεωρώ ότι η ανταλλαγή απόψεων είναι σημαντική δυνατότητα. Μπορώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου και για πρώτη φορά να συναντήσω τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών δραστηριοποιούνται στον τομέα δικαιοσύνη εσωτερικών, μεταναστευτικών πολιτικών και διαχείριση των συνόρων. Ξέρω ότι είναι κρίσιμο ο ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την υιοθέτηση ευρωπαϊκή νομοθεσία στου προαναφερθέντε τομεί. Ξέρω ότι είναι ρόλο του Κοινοβουλίου που αφορά δημοσιονομικά θέματα και γνωρίζω το βασικό ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο των φορέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό, υπό τη μελλοντική μου ιδιότητα, του εκτελεστικού διευθυντού του Frontex, θέλω να αναπτύξω καρποφόρες ε, σχέσεις με τα μέλη της Επιτροπής σας. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα συντομία να σας συστηθώ πριν να παρουσιάσω το πώς βλέπω τις προκλήσεις του Frontex στο μέλλον. Όπως θα γνωρίζετε πιθανότατα, Εργάστηκα επί 18 χρόνια σαν δημόσιος υπάλληλος στη Γαλλία, επίσης για τρία χρόνια στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για δύο χρόνια ήμουν διπλωμάτης στην Κορέα. Η καριέρα μου ε, εκινήθηκε μεταξύ στατηγικών και επιχειρησιακών προσεγγίσεων και μεταξύ εσωτερικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δραστηριοτήτων εκινήθηκα. Υπηρέτησα στο Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών το Υπουργείο Εσωτερικών στο Παρίσι, στο κέντρο του Υπουργείου που ασχολήθηκα με θέματα Σέγγεν και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, πολιτική θεωρήσεων, διαχείριση μετανάστευσης, σε τοπικούς, ε, σε τοπικά καταστήματα και σε ήμουνα ε, υπό αντινομάρχης. Ε, έπρεπε να ασχοληθώ σε τοπικό επίπεδο με ευρωπαϊκά θέματα, έπρεπε να συντονίσω διάφορους δημόσιους φορείς και δυνάμεις επιβολής της τάξης όπως αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Έχω συλλέξει πολλέ εμπειρίε, έχω περτήσει και σε άλλα υπουργεία και σε δημόσιε φορεί, στο Υπουργείο Άμυνα, στο Παρίσι, σαν επικεφαλή τη Διεύθυνση για Διεθνέ και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σαν ε, αντι, αναπληρωτής πρέσβης της πρεσβείας της Γαλλίας στην Κορέα και είχα αποσπαστεί σαν εθνικός εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Εσωτερικών από το 2000 μέχρι το 2003. Εκεί με, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσα να συμμετάσχω ενεργά συντάσσοντας την ανακοίνωση με τίτλο «Προς ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων» που εγκρίθηκε το 2002 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλης και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία ε, του Frontex. Ε, αυτή ήταν η εμπειρία που μου δημιούργησε φιλοδοξίες και ενδιαφέρον όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές δικαιοσύνης εσωτερικών και με έπεισε ότι θα έπρεπε να προσπαθήσω να υπηρετήσω ξανά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο μέλλον. Όπως βλέπετε, στις περισσότερες από τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησα, έμεθα πώς να γεφυρώνω το χάσμα μεταξύ στατηγικών προπτικών και συγκεκριμένης εφαρμογής στην πραγματική ε, ζωή, στην πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο όσον αφορά την επαγγελματική μου εμπειρία που θα ήθελα να παρουσιάσω διότι νομίζω ότι σχετίζεται με τις εργασίες Επιτροπής σας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω το πώς η Επιτροπή σας ασχολείται με το σεβασμό του κράτους δικαίου και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στις περισσότερες θέσεις τις οποίες υπηρέτησα, ελάμβανε υπόψη αυτές τις ανησυχίες. Ήταν ένα κομμάτι της αποστολής μου. Στην τελευταία μου θέση, στη Γαλλία, ήμουν σε στενή επαφή με φορείς που ασχολούνται με θεμελιώδη δικαιώματα και ήμουν σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που φρόντιζαν για τα δικαιώματα των μεταναστών. Στις διάφορες θέσεις μου ασχολήθηκα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έπρεπε να εφαρμόσω την αρχή της αναλογικότητας στα πλαίσια της ε, διαχείρισης των φορέων επιβολής του νόμου. Να δώσω περαιτέρω παραδείγματα συνέβαλα στη συνεργασία με διεθνή ε, ε, ποινική νομολογία και σε λιγότερο δραματικές περιστάσεις εργάστηκα στο Υπουργείο Αμήνης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σε ε, ειρηνευτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν το ιστορικό μου υπόβαθρο. Βεβαίως γνωρίζω, έχω πλήρη επίγνωση της Χάρτας Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η χάρτα που ισχύει και για το Frontex και θα εξασφαλίσω το ότι ο φορέας θα εφαρμόζει τις αρχές αυτές σωστά και θα τις προωθεί. Τώρα όσον αφορά τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Frontex τα επόμενα χρόνια, ε, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα στις αποστολές του οργανισμού και το όραμα που έχω για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει. Το, ο Frontex δημιουργήθηκε τόσο ώστε να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με μακροπρόθεσμη ε, προσέγγιση όσον αφορά τους επιχειρησιακούς και πολιτικούς στόχους, θεωρώ ότι ο Frontex θα διαδίδει έναν πολιτισμό εργασίας και το συνέστημα ότι όλα τα σύνορα πρέπει να τα, τα διαχειριζόμαστε μεζόμενες κοινέ αξίες. Ο Frontex είναι επιχειρησιακός φορέας που παρέχει την αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που είναι στην πρώτη γραμμή των εξωτερικών συνόρων. Ενώ παρέχει λοιπόν αλληλεγγύη, ο Frontex θα πρέπει παρόλα αυτά να μην ειδωθεί σαν ένας φορέας που θα υπερέχει των ευθυνών που έχουν τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Ε, για την ώρα θεωρώ ότι ο Frontex θα προωθεί όλο και ισχυρότερη σύγκληση μεταξύ των εθνικών φορέων των επιφορτισμένων με τη διαχείριση των συνόρων, έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον φορέα μας να εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τα σύνορα και για χρηματοδότηση του ελέγχου. Από, θεωρώ ότι είναι επιχειρησιακό τμήμα τη γενική προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά την κινητικότητα και τη μετανάστευση, που σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτύσσει ε, συνεργασία που δημιουργεί ε, δυνατότητε ε, σωστέ με τα τρίτα κράτη, με, με τρίτε χώρε. Θα συμβάλλει σε ευρύτερε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω ο Frontex και θεωρώ ότι ο Frontex θα είναι ένα φορέα που θα πρέπει να συνεργάζεται βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επιτόπου με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου, την, την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Europol, το SEPOL και το Eurojust. Ε, κυρίες και κύριοι, για να συνοψίσω τη βασική πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Frontex πολιτικές και επιχειρησιακές προσδοκίες είναι όλο και όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει να βρεθεί απάντηση όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση και θα πρέπει να υπάρχει και ψηλό επίπεδο όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Πολλαπλοί παράγοντες ίσως εξηγούν γιατί αυτό το θέμα τώρα είναι πλέον ορατό, πιο ορατό. Παρ' όλα αυτά οι, εκείνοι που χειρίζονται εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν πρέπει να υποτιμούν τις διαφορετικέ πίεσεις των δημογραφικών τάσεων και τη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική κατάσταση που επηρεάζει το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, οι μικτές ροές οικονομικών μεταναστών και ετούντων άσυλο προσπαθούν να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να, ε, να τα συμπεριλαμβάνουμε σε αποστολέ του Frontex και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των εκείνων που φυλάσσουν τα σύνορα. Και ούτω τρόπο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν επιχειρησιακά βήματα ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη επιβολή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως καθορίζονται από τον κώδικα του Σέγγεν για τα σύνορα. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό πιστεύω ότι ο ρόλος του Frontex είναι να δώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ε, έχοντας ευρύτερη εικόνα υπόψη. Λοιπόν, αυτή την ευρύτερη εικόνα, οι προκλήσεις για το Frontex θα μπορούν να κατανεμηθούν σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα επιχειρησιακής μορφής, οικονομικής μορφής ή ε, προβλήματα που αφορούν τη στελέχωση. Από πλευράς επιχειρησιακής τώρα, αν δούμε το θέμα το, ο Frontex θα πρέπει να πετύχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών επιλογών που υπάρχουν, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ροή μεικτών, ε, μεταναστών, ροών μεταναστών που διέρχονται τα θαλάσσια σύνορα Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς να αγνοούμε τα χερσαία σύνορα που ίσως και εκεί να ελοχεύουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι και απειλές, χωρίς να αγνοούμε τα αέρια σύνορα που ίσως να εκτίθενται σε παράτυπες μεταναστευτικέ ροές και απειλέ που προέρχονται πανταχώθεν. Ο οργανισμός επίσης θα πρέπει να πετύχει ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων κοινών επιχειρήσεων σε κατεπίγουσες καταστάσεις και μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε δημιουργία δυναμικού όπως το Eurosur ή θέματα κατάρτισης που θα έχουν στόχο ένα ευρωπαϊκό σύστημα για ε, ευρωπαίους μεθοριοφύλακες ο Frontex θα πρέπει να ασχοληθεί και με ένα παράδοξο που υπάρχει. Δηλαδή είναι επιχειρησιακός φορέας, αλλά εξαρτάται από του πόρου των κρατών μελών και το δυναμικό των κρατών μελών. Ε, ο φορέας λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσει τη θεσιμότητα των ε, στοιχείων των ε, μέσων των κρατών μελών μέσω της διαδικασίας pooling and sharing και ο φορέας θα πρέπει να βρει λύση το πώς να μισθώνει δυναμικό για περιόδους συγκεκριμένες αν χρειάζονται επιχειρήσεις για να βρεθούν γρήγορες απαντήσεις σε προβλήματα. Οικονομικός πώς. Ο Frontex έχει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και έχει γύρει ψηλέ προσδοκίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Και οι ψηλές αυτές προσδοκίες δημιουργούν μεγάλη πίεση στο Frontex. Μετά την αφετηρία και τις πρώτες χρονιές λειτουργίας θα μπορέσει και ο οργανισμός να αυξήσει το τμήμα των επιχειρησιακών δαπανών ε, έναντι των διοικητικών δαπανών. Εν πάση περιπτώσει, ο οργανισμός θα πρέπει να ετοιμάσει και την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και για κάτι τέτοιο θα πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες των στρατηγικών του δράσεων και ε, για να επιτύχει την υποστήριξη των ενδιαφερομένων αλλά και την ειδική υποστήριξη, μια και για τον προπολογισμό αρχή, θα πρέπει ε, να εκδώσει δημοσιονομικά δελτία που θα είναι ευανάγνωστα και διαφανή. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Οι προκλήσεις μας οφείλονται στις επιχειρησιακές και στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν ε, έχω ακόμη εμπειρία από τη λειτουργία του οργανισμού, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για τα διοικητικά θέματα και το προσωπικό. Ε, πάντως, κατά κανόνα, μέχρι τώρα θέλω να ε, ακούω τις απόψεις των εργαζομένων και να μπορέσω να δημιουργήσω η γνώμη για τις προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσωπικού. Πάντως ε, το προσωπικό του οργανισμού σε πολύ απαιτητικού καιρού ε, και σε χαλεπές ηθίκε επιτέλεσε πολύ αξιόλογο έργο. Από αυτή την άποψη θα φροντίσω ώστε να βρεθούμε και σε αυτήν την ενδιάμεση περίοδο σε κατάσταση πλήρης λειτουργία. Θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα κατανείμουμε το προσωπικό τις διάφορες προτεραιότητες και να βελτιστοποιήσουμε την αντιστοιχία μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων των ε, ε, εργαζομένων και των αναγκών και των αποστολών μας. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πιο ευέλικτο τρόπο εργασίας για να προσαρμοστούμε σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, θα ήθελα να επισημάνω τις εξή προτεραιότητες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την διαθεσιμότητα των ε, πόρων των κρατών μελών με βάση τη διαδικασία της κοινή συγκέντρωσης και διαχείρισης των πόρων, pooling and sharing. Επίσης να γίνει ε, ισόρροπη αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών συνόρων, χερσαίων, θαλάσσιων και σε κάποιο βαθμό και εναέριων. Επίση, κατά την προετοιμασία τη ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, θέλουμε κάποιου στόχου επιχειρησιακή συνεργασία με τρίτε χώρε, μη κοινοτικέ, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των συνόρων και την παράτυπη μετανάστευση, προκειμένου να ε, στηριχθεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κινητικότητα και την μετανάστευση. Κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι προκλήσεις ε, μας δημιουργούν ε, μεγάλες υποχρεώσεις. Είναι το έργο πολύ απαιτητικό. Έχω επίγνωση της ευθύνης και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Frontex. Η συλλογική προσπάθεια είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και προσβλέπω και στη δική σας υποστήριξη, γιατί κατά τη γνώμη μου η συλλογική προσπάθεια, το συλλογικό έργο είναι άρρηκτα δεμένο και με τη διαφάνεια. Οπότε σε αυτή την εποχή της διαφάνειας θα ήθελα να ξεκινήσουμε ανοιχτές και τακτικές σχέσεις μαζί σας. Οι επισκέψεις ε, στα κεντρικά γραφεία του Frontex έχουν ήδη προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο και θα ήθελα να σας απευθύνω και μόνιμη πρόσκληση σε όλα τα μέλη ε, της Επιτροπής που μπορούν να με επισκέφτονται όποτε θέλουν στη Βαρσοβία πέραν των επίσημων επισκέψεων αντιπροσωπιών της Επιτροπής σας. Επίσης, θα σας ε, ενημερώνω τακτικά για τις δραστηριότητες του Frontex και είμαι στη διάθεσή σας για ad hoc ενημέρωση σε περίπτωση ιδιαίτερων ε, συμβάντων ή ε, για θεματική ενημέρωση ανάλογα με τα θέματα που σας απασχολούν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, θερμά ευχαριστώ για την προσοχή σας. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νιγκέρη. Συνάδελφοι, δεν θα ακούσατε αυτά που θα είχα να πω στο τέλος της συνεδριάσεως, γιατί θα θέλετε να φύγετε όλοι προς το τέλος της συνεδριάσεως. Να πω ότι δεν έχουμε πολλά τέτοια θέματα την πέμπτη το απόγευμα. Να πω στους παρόντες συναδέλφους τώρα που είναι εδώ 4 και 10 και το προσωπικό ότι είναι καλό που είστε εδώ. Κάποιοι από εσά εργάζεστε σκληρά. Παρακαλώ συνεχίστε να είστε έτσι και το εκτιμούμε. Δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας στην Λίμπε με βάση το πρόγραμμά μας, αν δεν το κάνετε αυτό. Το εκτιμώ. Έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και αν δεν κάνουν τα μέλη αυτό που κάνατε σήμερα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και ευχαριστώ και το προσωπικό. Το λέω τώρα, διότι όταν τελειώσουμε το σημείο αυτό τη ημερήσια διάταξη, δεν θα με ακούσετε να τον τα λέω στο τέλο. Όταν φτάσουμε στα διάφορα, εσεί φεύγετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ποιοι είστε και εργάζεστε σκληρά και σας ευχαριστώ. Είναι καλό. Βέβαια, αλληλοσυγχαιρόμαστε. Είναι κάτι που κάνουμε σαν πολιτική. Κύριε Λογκέρη, είναι ασυνήθιστη αυτή η κατάσταση. Ε, είναι κάτι τυπικό που κάνουμε εδώ. Ε, καθορίζεται τις προτεραιότητες κλπ. Αλλά έτσι τα μέλη μας έχουν μια ευκαιρία να συζητήσουν προτεραιότητες κλπ. Υπάρχουν γνώσεις εδώ για το Frontex. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις Λοιπόν, να αρχίσουμε την κουβέντα μας, να αρχίσουμε τη διαδικασία, να σας υποβάλουμε ερωτήσεις και να συζητήσουμε τις ε, προτεραιότητες σας. Η Μπίρκετ είναι η πρώτη που... Η Μπίρκετ Σίπελ παίρνει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις θα μπορούσα να θέσω. Ο Frontex είναι ένας οργανισμός που συχνά συγκεντρώνει τα πειρά της κριτικής και καμιά φορά δικαίως γιατί μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα που κάνει. Καμιά φορά όμως και αδίκως, διότι καμιά φορά και χώρες μέλη δεν στηρίζουν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Μιλήσατε για στρατηγικά σημεία, κέντρα βάρους. Μιλήσατε και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Βλέπετε εκεί κάποιους συγκεκριμένους στόχους ενισχυμένη ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινέ δραστηριότητε. Τι μπορεί να εννοείται με αυτά. Εξάλλου, άλλο θέμα, πρόβλημα μάλλον, η διαφύλαξη των θεμελιωδών ελευθεριών. Είχαμε και μια έκθεση πρόσφατα για το τι συμβαίνει στα σύνορα, σε σημεία διαβάσεως των σύνορων και σε αεροδρόμια όπου δεν τηρούνται καμιά φορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Τι, γίνεται, τι χρειάζεται εκεί, χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση, χρειάζεται εσεί περισσότερο προσωπικό. Πού βλέπετε ότι πρέπει να ρίξετε το βάρος των προσπαθειών σας. Και μια τελευταία ερώτηση για τους χρηματοδοτικούς πόρου του, της λέει η κυρία Ζίπελ. Αν μπορούσατε να αποφασίσετε μόνο σας πού θα θέλατε να συγκεντρωθούν οι πόροι που διατίθεται για τον Frontex. Ευχαριστώ. Να πω ότι το Φεβρουάριο ετοιμάζουμε επίσκεψη επιτροπής μας στη, στον Frontex. Η Σεσίλια Βεκστρόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λετζέρη, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Λίμπε και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Πολύ σημαντική η θέση, το αξίωμά σας αυτό και προσβλέπουμε σε πολύ στενή συνεργασία. Πολύ ε, ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μου δώσετε από το βιογραφικό σας. Μα πότε ξεκινήσετε να υπηρετείτε στα κοινωτικά θεσμικά όργανα, από τον υπηαγωγείο. Όλα τέτοια, κάτι τέτοια λέει, μην την παίρνετε σοβαρά. Τα ίδια λέει σε όλους. Κλοντ, εγώ έχω το λόγο, μην με διακόπτεις. Όταν συζητήθηκε ο νέος κανονισμός για τον Frontex στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε ένα θέμα που επισημάνατε κι εσείς και τέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής και τότε και αποτελεί και η ψηφή μας προτεραιότητα ακόμη. Δηλαδή η εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Frontex. Και είπαμε ότι έχουμε και το συμβουλευτικό φόρουμ και ε, επεκτείναμε την κατάρτιση του προσωπικού του Frontex ε, και σε θέματα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και αν υπάρχει υπόνοια παραβίασης ε, θεμελιώδου δικαιώματο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της Frontex θα πρέπει ο ε, κατηγορούμενος υπάλληλος να, τεθείτε, να, να τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι ότου διαλευκανθεί η περίπτωση. Εσείς ως νέος εκτελεστικός διευθυντής του Frontex μπορείτε να διαβεβαιώσετε την Επιτροπή μας ότι θα εξασφαλίσετε σε κάθε περίπτωση σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τι μέτρα προβλέπετε σε περίπτωση παραβίασης από κάποιο υπάλληλο του Frontex αυτών των δικαιωμάτων. Πρόσφατα αντικαταστήσαμε την επιχείρηση Μάρε Νόστρου με την επιχείρηση Τρίτων. Εκεί είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δράσεων των κρατών μελών, προκειμένου της Ιταλίας με το Mare Nostrum και των δυνατοτήτων του Frontex σε σχέση με τον εξοπλισμό που έχει το μέγεθος των σκαφών και ούτω καθεξής. Θέλουμε ο Frontex να είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα μέσα και τους πόρους για να μπορεί και στα σύνορά μας και στην Μεσόγειο να ανταπεξέλθεται στο έργο του πριν τα τέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής αιτίας ε, λάβαμε την απόφαση για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις και ο σχετικός κανονισμός αναφέρει ότι η διάσωση ζώων είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Ελπίζω να μας ε, δίνετε συνεχείς αναφορές για το πεδίο εφαρμογής, για, την, για το βαθμό εφαρμογής αυτού του κανονισμού, για τις προβλεπόμενες ε, επιχειρήσεις και φυσικά τις δραστηριότητες από τη στιγμή που θα αρχίσει να εφαρμόζεται η επιχείρηση τρίτων. Ευχαριστώ και προσβλέπουμε σε συνέχιση των επαφών μας και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λεγκέρι, Λετζέρι, δεν ξέρω πώς είναι το σωστό. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεργασία που πλανάτε τώρα πάνω από το κοινό μας μέλλον και τη βρίσκω πολύ σημαντική μεταξύ Κοινοβουλίου και Frontex. Αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας σε δύσκολη περίοδο. Πολλές κρίσεις στη γειτονιά μας, υπάρχει και κρίση της μετανάστευσης και βεβαίως, α, βέβαια η χρηματοδότηση. Εξ αυτών απορρέουν δύο ερωτήματα. Πρώτο, σε ποια σημεία μπορεί το Κοινοβούλιο και ιδίω βεβαίως η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών να ενισχύσει την εργασία σας στο Frontex. Να ακούσουμε από εσά, δηλαδή τι είναι σημαντικό. Δεύτερο ερώτημα, προπολογισμό. Είναι σαφές ότι οι χώρες μέλη, μπορεί να πει κανείς, ότι εθελουσίως μάλλον δεν θα προσφέρουν περισσότερη χρηματοδότηση στον Frontex Υπάρχει όμως η αναγκαιότητα εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ιδιαίτερα να μην σιωπήσουμε στο μέλλον. Όταν δηλαδή το έργο σας υπονομεύεται από εκείνους που σας στερούν τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό και σας ρωτώ σε ποιο ύψο πρέπει να καθορίσουμε τον προπολογισμό. Από τη δική σα κοπιά, πόσα χρήματα χρειάζεστε. Um, Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Ο κύριος Σιρόφσκι, Τόμας. Καλύτερα το είπα τώρα. Ναι, καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κλοντ, είσαι έξοχος. Γίνεσαι σαν τη Σεσίλια. Υπερβάλλεις τώρα, υπερβάλλεις. Άκουσε στα τσεχικά και βλέπω ότι τώρα έχεις καλύτερη προφορά. Ξαναγύρισέ το στα τσεχικά. Θα μιλήσω τσεχικά. Θα σας πω λοιπόν, κύριε Λετζέρη, ε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ που ε, έχετε ανοιχτό πνεύμα και είπατε ότι μπορούμε να έρθουμε να σας επισκεφτούμε και πράγματι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι και τόσο μακριά. Κυρίως από την Πράγα, από την Τσεχική Δημοκρατία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για την επίσκεψή μας. Αλλά θα έχουμε και σκληρές ερωτήσεις να σας θέσουμε. Είμαι εισηγητής ή μάλλον σκιώδης εισηγητής για το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι αυτό το Ταμείο κατά το παρελθόν δεν συμμετείχε πολύ στις επιχειρήσεις Frontex και ε, οι πόροι των κρατών μελών δεν διατίθενται στο Frontex. Πώς θα αλλάξετε την κατάσταση, έχετε κάτι υπόψη σας. Δεύτερον, στο βιογραφικό σας αναφέρετε ότι έχει μεγάλη εμπειρία για εργαζόμενος για πολλά θεσμικά όργανα και διοικήσεις. Έχουμε εμπειρία με ανθρώπους που είναι ε, δημόσιοι υπάλληλοι που θεωρούν ότι τα πράγματα μπορούν, ε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Ελπίζω ότι, ότι στο Frontex θα εστιαστείτε επιβελτιώσεως ε, των εργασιών. Ήμουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό φέτος και το 2015 και στην πρόταση του Συμβουλίου διαπίστωσα ότι αναμένεται περικοπή των πόρων που διατίθενται σε εσάς ίσως να περικοπεί και το προσωπικό σας. Αυτό πώς σας επηρεάσει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά. Όπως και η Σεσίλια, θέλω να επενέσω και την διερμηνία. Πριν μιλούσα γερμανικά και άκουγα την τσεχική διερμηνία, ήταν τέλεια η διερμηνία. Νομίζω καμιά φορά θα πρέπει να επενούμε και τους διερμηνείς μας για την καλή δουλειά που κάνουν. Συμφωνώ πολύ. Θεωρούνται σαν κάτι δεδομένο. Συμφωνώ. Ευχαριστώ, Τόμας. Η κυρία Μέιερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Λετζέρη για την παρουσία του στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε παρόντες για να ακούσουμε τον κύριο Λετζέρη. Ο οργανισμός Frontex ε, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας με όλες αυτές τις ροές μεταναστών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προσέξουμε την οργάνωση του Frontex. Πιστεύετε ότι ε, επί της δικής σας θητείας θα δώσει ο Frontex μια λύση στην μετανάστευση, στην νόμιμη μετανάστευση. Πώς θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Θα μπορέσουμε να σταματάμε τους παράτυπους μετανάστες στα σύνορα. Äh, Έχω μια ερώτηση. Μιλήσατε και για τη συνεργασία σας με Ευρωπολ, Eurojust κλπ. Σχεδιάζεται συμφωνία. Αυτό θέλω να μάθω. Κατά πόσο έχει προχωρήσει για την ανταλλαγή δεδομένων, η συμφωνία αυτή δηλαδή, μεταξύ Frontex, Europol, Eurojust κτλ. Στην αρχική σας ομιλία εξηγήσατε ότι θεωρείτε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως πολύ σημαντική και ότι έχετε και σχετική εμπειρία. Κύριος Ράντεφ, επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λετζέρη, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για το διορισμό σας στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Frontex. Αναλαμβάνετε τη θέση σας ε, σε μια εποχή υψηλών προσδοκιών απέναντι στο Frontex, γιατί ο Frontex καλείται να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα από την παράτυπη μετανάστευση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει προστασία στους ετούντες άσυλο. Ως Ευρωβουλευτής από τη Βουλγαρία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερος για τους ε, αιτούντες άσυλο γιατί ε, η Βουλγαρία δέχεται πολλούς ε, σύρους αιτούντες άσυλο, σύρους πρόσφυγες. Πάνω από 30.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν παράνομα τα βουλγαρικά σύνορα φέτος μόνο. και μάλιστα μερικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην Βουλγαρία από την Μαύρη Θάλασσα. Ζητήσαμε βοήθεια από τους ε, Ευρωπαίους συναδέλφους. Ερωτώ λοιπόν, θα πραγματοποιήσετε αποστολή στη Βουλγαρία, κυρίως στα βουλγαροτουρκικά σύνορα και στα βουλγαροελληνικά σύνορα γιατί πιστεύω ότι θα χρειαστούμε αποστολή και επιχείρηση του Frontex και στον Εύξηνο Πόντο για να περιορίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Μήπως ε, και θα, η Μαύρη Θάλασσα, ο αυξηνος Πόντος θα γίνει νέα διάβλος εισόδου ε, μεταναστών και προσφύγων μετά τη Μεσόγειο. Επίσης, ποια είναι τα μακροπρόθεσμα μέτρα σας για χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται συμπληρωματική βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τι τεράστιε μεταναστευτικέ ροέ. Ευχαριστώ κυρία Έλλη Σλάιν. Ε, Ευχαριστώ, σα καλωσορίζω και εγώ. Έχω μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη για σα. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε το ρόλο του οργανισμού Frontex όσον αφορά την επιχείρηση τρίτων. Από τον Οκτώβριο του 2013, από την τραγωδία της Λαμπεντούσα, η Ιταλική κυβέρνηση ε, ξεκίνησε την επιχείρηση Mare Nostrum που κατάφερε να διασώσει πάνω από 100.000 ε, ζωές στη Μεσόγειο που δυστυχώς η Μεσόγειος όπως είπε κάποιος έγινε ένα κημητήριο ευρωπαϊκό καταφέραμε να κάνουμε πρώτα ένα ευρωπαϊκό κημητήριο πριν έχουμε πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Αυτή είναι η τραγωδία. Είναι θετικό ότι υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση που συντονίζει ο Frontex και συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη που ασχοληθεί τη σωστή ε, προσέγγιση να αντιμετωπίσει την πρόκληση μετανάστευση σαν ευρωπαϊκή ε, πρόκληση που δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη που είναι στα σύνορα, τα νότια σύνορα της Ευρώπης. Όμω υπάρχουν και πάρα πολλέ ανησυχίε, διότι από τη μία πλευρά τα διαθέσιμα μέσα για το τρίτον, όπω είπε και η προλαλή σα ε, η κυρία Βίξτρομ, ε, δεν μπορούν να συγκριθούν καν με εκείνα που έχουν ε, διατεθεί για το Μαρενόστομ. Λιγότερα αεροσκάφη, λιγότερα σκάφη και λιγότεροι άνθρωποι, λιγότερο προσωπικά. Η περιοχή της παρέμβασης δεν είναι στα 172 από τα χωρικά υδάτα, αλλά μόνο στα 30 μίλια. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο. Και τέλος γιατί δεν είναι σαφό αν το τρίτον θα έχει μια εντολή για έρευνα και διάσωση όπως είχε το Μαρενόστρομ. Πιστεύω λοιπόν ότι μειώνοντα την ακτίνα τη παρέμβασή μα θα δούμε νέε τραγωδίε, πιστεύω, ή χειρότερα να μην τι βλέπουμε, όπω συνέβαινε πριν να έχουμε μια επιχείρηση ε, με τα σκάφη εκεί. Θα σα ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλο ε, του Frontex στην επιχείρηση τρίτων, τι σκέφτεσαι για αυτέ τι ανησυχίε όσον αφορά τη λειτουργία αυτή και πώς μπορεί να ενισχυθεί ενδεχομένως η αποστολή αυτή. Αυτό να τους. Όπως ξέρετε κάποια από τα μέλη μας έχουν πάει εκεί. Έχουν πάει επί τόπου. Εδώ είναι αυτή η εμπειρία πολλών μελών της Επιτροπής μας. Είναι πολύ περίπλοκες ερωτήσεις, έξοχες ερωτήσεις και περιμένουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Παρακαλώ προς, εάν μπορείτε να απαντήσετε όσο πιο λεπτομερώς μπορείτε, αλλά και σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη. Ορίστε, έχετε το λόγο. Well, uh, thank you. Σας ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ για την πληθώρα των ερωτήσεων. Θα μιλήσω τώρα γαλλικά και προειδοποιώ τους διερμηνείς. Bien, je... Πολλές ε, ερωτήσεις αφορούσαν τα δημοσιονομικά θέματα και τη χρηματοδότηση. Γνωρίζετε ότι ο προπολογισμό του 2014 για το Frontex ήταν 90 ε, εκατομμύρια ευρώ. και έγινε μια πρόταση για το αποθεματικό των 20 εκατομμύριων. Μακροπρόθεσμα και εννοώ εδώ το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιτελέσουμε με ακρίβεια το έργο μας ή δυνατόν ε, σε αγαστή συνεργασία με τους περισσότερους ε, φορείς και πέραν της συνεργασίας που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουμε συναντήσεις και συζητήσεις και με τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προπολογισμό αρχής και φυσικά δηλαδή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα, μια και διανύουμε χαλεπούς δημοσιονομικούς καιρού και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων του οργανισμού μας. Θα πρέπει να δικαιολογήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την αποτελεσματικότητα των επιλογών μας και να πιάνουν τόπο τα χρήματα που αφιερώνονται στο Frontex και τηρούμε αποτελεσματικά το έργο μας, αντιμετωπίζοντας και τις ανθρωπιστικές προκλήσεις, αλλά και την πρόκληση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Γιατί αυτή είναι η πρωταρχική αποστολή του οργανισμού Frontex. Τώρα, ως προς τα δημοσιονομικά θέματα, φυσικά θα θέλαμε την υποστήριξη της Επιτροπής σας. Θα ήταν πολύτιμο για μας κάτι τέτοιο και ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές που με ρώτησαν πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να βοηθήσει τον Frontex. Και θα χαρούμε ιδιαίτερα αν μας υποστηρίξετε κατά την αναθεώρηση που σχεδιάζουμε του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Προς το παρόν πάντως δεν μπορώ να δώσω ακριβείς προβλέψεις για τις χρηματοοικονομικές μας ανάγκες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακόμη δεν έχω αναλάβει επίσημα τα καθηκοντά μου. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω εδώ ένα νούμερο στην τύχη. Έχουμε όμως ε, και κάποιες ε, στρατηγικές προτεραιότητες που θα πρέπει να τις καθορίσουμε από κοινού με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του Frontex αλλά και σε συζητήσεις που θα γίνουν σε άλλα φόρα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα όλα τα θεσμικά όργανα θα συμβάλλουν με τις ενδείξεις τους και τις κατευθυντήριες τους γραμμές στην διαμόρφωση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στην ιεράρχησή τους. Και μετά από τέτοιες συζητήσεις και με βάση όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να δώσουμε με ακρίβεια ένα νούμερο για τις ε, χρηματοοικονομικές μας ανάγκες. Επίσης, ε, τέθηκαν ερωτήσεις για τη χρήση των ε, κοινοτικών κονδυλίων αν κατάλαβα καλά. Από το 2014 έχουμε τη νέα γενιά των ταμείων. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Ταμείο ε, της Οικογένειας, ΕΜΙΦ, τα αρχικά του στα αγγλικά. Και έχω την αίσθηση ότι ο Frontex μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να καταθέσουν επιλέξιμα σχέδια στα ευρωπαϊκά ταμεία και μπορούμε με την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωσία μας να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη ώστε να υποβάλουν ε, αιτήσει για επιλέξιμα προγράμματα και στη συνέχεια ο οργανισμός μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για κοινή χρήση των μέσων, κυρίως των επιχειρησιακών μέσων, των ε, πιο βαριών όπως είναι αεροσκάφη και σκάφη και που θα μπορούν να τα αγοράσουν κράτη ή ομάδες κρατών και που θα με βάση το pool and sharing θα τα χρησιμοποιούν από κοινού. Οπότε ο οργανισμός Frontex μπορεί να ετοιμάζει το πρόγραμμα και κυρίως να οργανώνει αυτή την κοινή συγκέντρωση και κοινή διαχείριση των πόρων, το pooling and sharing, διοργανώνοντας και κοινέ ομάδες περιπολίας σε περιφερειακό επίπεδο και με συμμετοχή πολλών κρατών μελών. Il y a plusieurs questions qui se sont exprimées. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για τον τρόπο προαγωγής τους και εφαρμογής τους. Είναι όντως σημαντική αυτή η αποστολή που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια Frontex. Έχουμε ειδικό υπάλληλο, επόπτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία ότι είμαι απόλυτα αποφασισμένος για να λειτουργήσει εύρυθμα αυτό το σύστημα σωστής εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, έχω δεσμευτεί για πλήρη σεβασμό του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε επιτόπου βέβαια τι συμβαίνει θα γίνονται τακτικές αναφορές, γιατί μπορεί να έχουμε συστήματα που γενικά και στη θεωρία είναι καλά οργανωμένα για το σεβασμό και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά μπορεί να έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων υπαλλήλων που για τον ΑΒ λόγο είτε παραβιάζουν είτε παρουσιάζουν κάποιες παραλήψεις στην άσκηση των καθηκόντων τους. Αλλά θα γίνει περιπτωσιολογική ανάλυση των υποθέσεων αυτών. Τέθηκαν ερωτήσεις και για τα ανατολικά σύνορα της Μαύρης Θάλασσας ή τα χερσαία σύνορα με μαζική εισρωή ετών τον άσυλο στη Βουλγαρία. Είπα και στην αρχή ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ταυτόχρονα με την βασική μας προτεραιότητα που είναι η κατεπίγουσα διαχείριση των θαλασσίων νοτίων συνόρων μας, αλλά ταυτόχρονα να μην αμελούμε την ανατολική πλευρά. Και θα πρέπει να δούμε με τα δημοσιονομικά μέσα που θα έχουμε, τι επενδύσεις θα κάνουμε στο μέλλον, πού θα επικεντρώσουμε τις ικανότητές μας και τι είδους επιχείρηση θα αναλάβουμε. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την βοήθεια των κρατών μελών στο Frontex και σε χώρες που σήμερα δεν έχουν επιχειρήσει Frontex, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους συνοριοφύλακες ε, των κρατών μελών. Δεν ξέρω. Από τώρα δεν μπορώ να σας βεβαιώσω ότι θα γίνει κάποια αποστολή στη Βουλγαρία, αλλά σίγουρα θα μεριμνήσουμε για να μην ε, παραμελήσουμε κανένα σύνορο και να μπορούμε να πάσα στιγμή να αναπτύσσουμε τις αποστολές μας και τους ε, υπαλλήλους μας όπου χρειάζεται χωρίς να επικεντρώνει την προσοχή μας μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε επανειλημμένως το θέμα της ικανότητας του Frontex να ελέγξει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα. Μην ξεχνάτε ότι με βάση τις συνθήκες τα κράτη είναι πρωτίστως υπεύθυνα, τα κράτη-μέλη και ο Frontex επεμβαίνει από έτσι των κρατών μελών για να επιφέρει μια προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή και την επιχειρησιακή του ικανότητα. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός Frontex είναι ένα ψηφιδωτό μόνο σε ένα ευρύτερο πλέγμα διατάξεων για την μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θα συνδράμει επιχειρησιακά ο Frontex στη διαχείριση των συνόρων αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα των χωρών προέλευσης ε, της παράτυπης μετανάστευσης, των χωρών διαμετακόμισης, διέλευσης και να αναπτύξουμε προγράμματα συνεργασίας, ε, αναπτυξιακής βοήθειας, ε, βοήθειας αποκατάστασης ή ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Υπάρχει μια σειρά πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί μακροπρόθεσμα να αποφέρει καρπούς και στον τομέα αυτό. Οπότε ο Frontex, ο οργανισμός μας, δεν είναι ο μόνος μηχανισμός ε, που έχουμε για να λύσουμε τα προβλήματα στις μεταναστευτικές ροές. Αναφέρθηκε και η επιχείρηση τρίτων και ο ρόλος του Frontex στη νέα αυτή επιχείρηση. Δεν έχω αναλάβει ακόμα, όπως σας είπα, τα καθήκοντά μου. Οπότε δεν είμαι ακόμη πλήρως κατατοπισμένος για την κατάσταση και το ρόλο του Frontex ε, στην νέα επιχείρηση. Ξέρω ότι είχαμε 47 περιπτώσεις, τουλάχιστον χθες 47 ήταν οι περιπτώσεις ε, στις οποίες ε, βοηθήσαμε με βάση την επιχείρηση Frontex και σώσαμε 47 ανθρώπους που κινδύνευαν να πνιγούν. Η εντολή της επιχείρησης τρίτων διαφέρει από την προηγούμενη Ιταλική επιχείρηση Mare Nostrum που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2003 με πρωτοβουλία της Ιταλικής κυβέρνησης και μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα. 2013, συγγνώμη. Και φυσικά, όπως, σας όπως είπατε κι εσείς, η επιχείρηση τρίτων είναι διαφορετικά πως πιο περιορισμένη. Ο ρόλος του Frontex πάντως είναι να αποφύγει θανάτους να αποφύγει να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους. Και όλοι όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση, όποια και είναι η αποστολή τους, όλα τα σκάφη που πλέον εκεί κοντά οφείλουν να παράσχουν βοήθεια. Αυτό προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Όλοι έχουν υποχρέωση παροχής βοήθειας και τα σκάφη του Frontex επίσης οφείλουν να εφαρμόσουν το δίκαιο της θάλασσας που δεσμεύει όλα τα κρατη και φυσικά και τον οργανισμό μας. Είναι ανθρωπιστική υποχρέωση και καθήκον η διάσωση ζώων. Αυτά προς το παρόν. Διότι δεν έχω αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά μου. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Είμαι στη διάθεσή σας βέβαια κυρίες και κύριοι βουλευτές για άλλες ερωτήσεις αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Λετζέρη. Όταν αναλάβετε τα καθήκοντά σας θα έχουμε ενδελεχέστερη συζήτηση. Για τα επιχειρησιακά ζητήματα θα είσαστε στην πρώτη γραμμή και θα έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση των θεμάτων. Θα σας επισκεφτούμε το Φεβρουάριο, οπότε θα μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος, θα μπορούσατε να είστε πιο αναλυτικός, το ξέρω αλλά θα έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Ευχαριστώ τα μέλη που ε, πήραν το χρόνο να μείνουν εδώ και νομίζω ότι θα διαπίστωσαν ότι άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ συνάδελφοι που μείνατε και έτσι άξιζε τον κόπο και η συζήτηση. ευχαριστώ και το προσωπικό για τη σκληρή δουλειά που έκανα την εβδομάδα και τους διερμηνείς. Ε, καλό Σαββατοκύριακο συνάδελφοι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.